Αυτή την απόφαση λοιπόν την μεταβίβασα στην αρμόδια Ιταλική Αρχή. Επίσης από το ομάδε του ΕΛΚ και του ΙΕΦΤΗ έλαβα πολλέ ε, αιτήσει για αλλαγέ σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και αντιπροσωπείε και ο κατάλογος των διορισμών θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει και δεν επιβληθούν παρατηρήσει ω την έγκριση των πρακτικών, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν εγκεκριμένοι. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στι αύριο, στι 22 Οκτωβρίου 2009, από